κείμενο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Λοιπόν. Και η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης. Για το χρονοδιάγραμμα εργασιών των Συνόδων Ολεμελίας έλαβε απόφαση διάσκεψη των Προέδρων την 5η 30 Απριλίου. Ε, πρόκειται για το χρονοδιάγραμμα εργασιών του 2016. Έχετε τις σχετικές ημερομηνίε στην ιστοσελίδα και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών